So. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η διάσκεψη των Προέδρων μόλις αποφάσισε για την απονομή του πραμίου Ζαχαρόφ του Νάντια Μπασάε και Λαμίγια Ζιμπασάρ. Κυρίες και κύριοι, η Νάντια Μουράτ Μπασάη και η Λαμίγια Ζιμπασάρ. Μπασάρ